και ο πρόεδρος ε, ρωτά τους διερμηνείς κατά πόσον ε, λειτουργεί τεχνικά ο ήχος. Ο ήχος λειτουργεί. Για την ελληνική καμπίνα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κηρύσω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 23 Ιουνίου σε απόλυτη συμφωνία με τις ε, πολιτικέ ομάδες συγκάλεσε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση δυνάμει του άρθρου 146 παράγραφος 4 υπό παράγραφο 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δοθεί η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να συζητήσει για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που συγκαλείται τόσο βραχυπρόθεσμα μία ολομέλεια. Αυτό λοιπόν το έκτακτο μέτρο είναι η αντίδραση και σε ένα μοναδικό γεγονός, χωρίς προηγούμενο, το γεγονός δηλαδή ότι ένα κράτος μέλος αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω το γεγονός ότι το σύνολο του σώματος των επιτρόπων βρίσκονται σήμερα κοντά μας συμπεριλαμβανομένου και του Επιτρόπου Χίλ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά σε αυτή την έκτακτη ολομέλεια. θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στο Κοινοβούλιο, στο λίκνο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ε, να διεξάγουμε μια συζήτηση για ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους και μάλιστα πάρα πολύ. Διότι κυρίες και κύριοι, σε αντίθεση με το σχολιασμό που έχει γίνει σε κάποια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση που ελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια απόφαση του Βρετανικού λαού και είναι μια απόφαση η οποία όμως αγγίζει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα οι ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σήμερα για το θέμα αυτό. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση, επιτρέψτε μου να δηλώσω τα εξής. Για τέσσερις ολόκληρες δεκαετίες, πολλοί πολιτικοί και κυρίως πάρα πολλοί υπάλληλοι Πάρα πολλοί λοιπόν μετέβησαν και εργάστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εγώ προσωπικά για όλες αυτές τις δεκαετίες συνεργάστηκα με συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο και προσπαθήσαμε από κοινού να οικοδομήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γι' αυτό λοιπόν και θεωρώ ότι ομιλώ και εξ ονόματός θεωρώ ότι μπορώ να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς τους συναντέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλους αυτούς τους άγνωστους εκατοντάδες άντρες και γυναίκες οι οποίες εργάστηκαν από κοινού με εμάς για την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μου να πω ότι λυπούμεθα βαθύτατα για την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας να θελήσει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σε εσά συνάδελφοι που συνεργαστήκατε μαζί μας νιώθουμε ότι πρέπει να σας εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά την αξία του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως στην εξωτερική πολιτική της Ευρώπης, αλλά και στην προάσπιση των ελευθεριών το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Από την άλλη όμως πρέπει να γίνει σεβαστή και να ενεργοποιηθεί η βούληση, η ετοιμιγορία του Βρετανικού λαού. Γι' αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα εντελεχώς και σε βάθος για την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω κάποιον που παρίσταται στην αίθουσα, κάποιον ο οποίος κατά τη γνώμη μου σε πολύ δυσχερείς συνθήκες εργάστηκε σκληρά, ιδιαίτερα αποδοτικά και έκανε ένα πολύ σημαντικό προσωπικό βήμα. Ο Λόρδος Χιλ δέχτηκε τις συνέπειες της στάσης του ως Επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα λοιπόν ο Λόρδος Χίλ είναι τελευταία φορά κοντά μας και πρέπει να σας πω Λόρδε Χίλ ότι εργαστήκατε για την εκστρατεία του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα αυτά που προσφέρατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.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 σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ και σας για το μήνυμα που εκπέμψατε και που δείχνει ποια ακριβώς είναι η στάση της δρυπτικής πλειοψηφίας των ευρωβουλευτών. Είναι στο πλευρό εκείνων που επιθυμούν ή επιθυμούσαν να διατηρήσουν την Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα βέβαια είναι απόλυτα σαφές ότι η παρέτηση του Λόρδου Χιλ είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός το οποίο έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις. Έχει φτάσει λοιπόν στιγμή, κυρίε και κύριοι, στιγμή για να συζητήσουμε και το λόγο έχει εκ μέρου του Συμβουλίου ο εκπρόσωπος ε, της Ολλανδικής ε, Προεδρίας, Χανή ε, Πλεσά. Και κυρία Χανή Πλεσά, εμείς νιώθουμε ιδιαίτερο σεβασμό για σας που εκπροσωπείτε